So Λοιπόν, προσπαθούμε ε, για μια δεύτερη φορά. Καλώς ορίσατε όλοι. Νομίζω ότι θα περάσουμε την ημέρα ψηφίζοντας. Και ελπίζω ως πρόεδρος ε, να μην σας απογοητεύσω, γιατί είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε ζητώ ήδη συγγνώμη σε περίπτωση που κάνω κάποιο λάθος. Για κάποιους συναδέλφους είναι επίσης η πρώτη φορά γιατί είναι νέοι, οπότε καλώς ορίσατε όλοι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απαλλαγή του 2018. Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ω εισηγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μου εισηγητέ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ όλους για τις εξαιρετικές συνεδριάσεις κοιοδών και τις πολύ καλές συνομιλίες ε, με τους συμβούλους και τους βοηθούς μας και ριτά, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία γιατί δεν είναι πάντα εύκολο όταν είναι όλοι νέοι και τα πάντα τα κάνουν για πρώτη φορά και ξεκινούν από το μηδέν. Και έτσι ελπίζουμε τώρα να η ψηφοφορία να πάει μια χαρά. Do it in the English language. Θα κάνουμε την ψηφοφορία στα αγγλικά γιατί μερικές φορές η μετάφραση αργεί. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω στα αγγλικά και ελπίζω να λειτουργήσει καλύτερα για όλους. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 1 του κυρίου Φλάναγκαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 Καταπέπτει. Τροπολογία 3 υπέρ. Α, συγγνώμη. Πρώτα χρειάζεται να έχω τον κατάλογο ονομαστική ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε, ποιος ψηφίζει υπέρ της απαλλαγής, ε, υπέρ. Είναι η τελική ψηφοφορία για την πρόταση για απόφαση για απαλλαγή της Επιτροπής. Ποιος δεκατά, αποχές. Ονομαστική ψηφοφορία είναι. Be... Είναι η πρώτη μου, ε. Θα τα πάω πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Λοιπόν, αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. <laughs> vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 20. Adopted 20 in favor εγκρίνεται 20 υπέρ και 4 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Τώρα περνάμε στην πρόταση της απαλλαγής. Α, δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε όλες. Απλά μπορούμε να πάμε στη σελίδα 5, στο σημείο 9 για την πρόταση ψηφίσματος, γιατί άμα ψηφίσουμε αυτό, περιλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, Πάμε στη συμβαστική 1. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 17, 18, 19, 16 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22, 21, 57 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 27. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβιβαστική 4 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην συμβιβαστική τώρα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στη συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην ε, συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 43 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 με προφορική τροπολογία υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία όχι με την προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 51. Ονομαστική ψηφοφορία, ποιο είναι υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το email δεν έφτασε και γι' αυτό είναι το υπάρχει πρόβλημα. This is as, I, as chair I can do it. Ως πρόεδρος ε, αυτό έκανα εγώ στο πρωί everybody could do roll call for them, but nobody asked them. Ονομαστικές ψηφοφορίες δεν τις ζήτησε κανένας. But I uh, don't think this is a big problem. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. That's a decision at the moment of the chair, but... Είναι απόφαση του Προέδρου τώρα αυτό, αλλά το ζήτησαν κιόλας. Ωραία να ελέγξουμε. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται πέρας ψηφοφορίας. «22 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή». Συμβιβαστική 12. Είναι ονομαστική επίσης η 12. Α, όχι, αυτή είναι η τροπολογία 52 μάλιστα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Μόνο έξι είναι οι ονομαστικές ψηφοφορίες. Για τη συμβιβαστική 12 άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 18 κατά τρεις, ε, τέσσερις αποχές. Τροπολογία 56 Φων Κράμον με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση. Όχι. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. 54. Έχουμε έξι ονομαστικές, το είπα. Λοιπόν, 23, 24, 24, 25 και 50. Εκεί ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία από το ΕΛΚΑ. 54 είναι ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ 0 αποχές 0 κατά 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές θα την ελέγξουμε Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 59. 59. Πέρας. Απορρίπτεται με 16 προς 10. Πάμε στη συμβιβαστική 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61-63 καταπίπτουν Θέλετε να ελέγξετε την 60 Ωραία, σε ελέγξουμε την 60 Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίφθηκε 12 με 10 και 4 εποχές. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται νομίζω. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν θέλετε, ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. «62 ψηφίζουμε». Ελέγχουμε την 62. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 με 10. 64. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 66 είναι στη συμβαστική 24 μαζί με την 68. Οπότε πάμε στην 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, δεν γίνεται ψηφοφορία για την 69. Ποιο είναι υπέρ. 69. Δεν γίνεται ψηφοφορία για την 65. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Είναι ευκολότερο. Vote is open. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται 14, 5, 7 αποχές 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ερέξουμε, Νομίζω ότι εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να μας λέτε τι τσεκάρουμε όταν το ελέγχουμε, είναι ευκολότερο για όλου. Το είπα, 74 λέει ο πρόεδρο. 74 είπα και μετά είπα να ελέγξουμε την 74. Ελέγχουμε την 74, ονομαστική. Εγκρίνεται με 16, 9 κατά και μία αποχή. 75 κατά πίπτη, συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 και 77 καταπίπτουν 78 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά έχουμε την 79 με προφορική τροπολογία ε, κάποιος που έχει ένσταση προς την προφορική τροπολογία όχι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 και 83 καταπίπτουν 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να το ελέγξουμε την 88 88 να άνοιξει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας 18 ως προς 8 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92, 91 κατά πίπτουν, 94 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία 93 έτσι 93 ψηφίσμα. πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 11. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι να το παληθεύσουμε μια στιγμή ψηφίζουμε επί του 100 εγκρίνεται το 100 νομίζω 100 ψηφίζουμε έγινε ένα λάθος έτσι για το 100 ψηφίζουμε λοιπόν Άρχεται ψηφοφορία για το 100. Πέρας ψηφοφορίας. Νομίζω εγκρίνεται. Ναι, ναι, εγκρίνεται. 98. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99. Εδώ έχει, έχουμε μια αλλαγή στην ημερομηνία. Προφορική τροπολογία, δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση. Υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. 101. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, Συμβασμό 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 και 209 καταπίπτουν. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105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 Συμβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 113 και 112 καταπίπτουν. Συμβασμός 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 και 114 καταπίπτουν. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 με προφορικές τροπολογίες υπάρχει αντίρρηση όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 125 να επαληθεύσουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία για το 125 πέρας ψηφοφορίας 15-10 απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά εδώ θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό νομίζω άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 13-12 εγκρίνεται και τώρα 128 υπέρ κατά πάλι θα πρέπει να παληθεύσουμε για το 128 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 13-10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 αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω να το επαληθεύσουμε ποιος είναι υπέρ μάλλον άρχιτη ψηφοφορία συγγνώμη άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 137 έτσι εγκρίνεται 16.8 142 υπέρ κατά νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία πάλι εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 με προφορική τροπολογία υπάρχει αντίρρηση όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις υπέρ κατά είμαι η ε, να το επαληθεύσουμε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 Πινιεντόλη 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε 155-156 καταπίπτουν και πάμε στην 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 προφορική τροπολογία υπάρχει αντίρρηση όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 23 ορματική ψηφοφορία παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 23 με τρεις αποχές, 23 με αποχές οι άλλες τροπολογίες εδώ καταπίπτουν και πάμε στην συμβαστική 24 ενωμαστική ψηφοφορια ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 22-3 και τώρα πάμε στον συμβιβασμό 25 και πάλι ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται 19 και 4 εποχές και 2 ψήφοι κατά. Πάμε τώρα στην 177 υπέρ ...178 τελικά... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...179... Όχι, απορρίπτεται, συγγνώμη, απορρίπτεται, δικό μου το λάθος. Λάθος λέξη. 179, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει. Συγγνώμη, έχω ένα ερώτημα. 178 καταπίπτει. Έτσι δεν είναι. Όχι, απορρίφθηκε το 178. 178 ζητούσε να διαγραφεί όλη η παράγραφος, δεν ήταν μέρος του συμβασμού. Ψηφίσαμε και πριν 179, 180 καταπίπτει, μια και ψηφίσαμε υπέρ στην 179 και πάμε στο συμβασμό 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 182 καταπίπτουν και πάμε στην συμβασμό 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν 184 185 183 πάμε στην 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά ναι. αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι απορρίπτεται ναι ναι αυτόματα τα λέω 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 προφορική τροπολογία έχει κάνει αντίρρηση όχι ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εξήνεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 η νέα ψηφοφορία. Δεν, είπα, δεν ψηφίζουμε εδώ γιατί είναι συγγνώμη γλωσσική τροπολογία. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 δεν ψηφίζουμε. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε αυτό 204 άρχιτη ψηφοφορία We close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας 12 προς 11 εγκρίνεται. 205 με προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, δεν βλέπω κανέναν. We are in 205 ε, υπέρ. Με την προφορική τροπολογία είναι συν. 205 υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. 206 καταπίπτει, 207 με προφορική τροπολογία, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, εδώ πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το 2008. We close the vote. 13-11 ε, εγκρίνεται. 209 είναι μέρος της συμβαστικής λύσης 18. 210. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε. 210. 210. Επαληθεύουμε. Α, αποσύρεται. Α, αποσύρεται. Εντάξει. Ε, 210 αποσύρθηκε λοιπόν. 211 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 213, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 214, υπέρ, είναι συμβατές, δεν είναι. Η 14, 214. Ψηφίζουμε για την 214. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215, τώρα καταπίπτει. 216, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 217, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 218, μάλιστα. Να το επαληθεύσουμε για το 217 λέτε. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλετε ε, ονομαστική ψηφοφορία για την 218 λοιπόν. 218. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 προς 7. 219. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 220. Υπέρ, κατά, Ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 220. Πέρας της ψηφοφορίας. Σαφώς απορρίπτεται με 17 ψήφους. Μετά πάμε στην 222. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225, υπάρχει προφορική τροπολογία εδώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 226, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 228, υπέρ, κατά, ας το επαληθεύσουμε στα γρήγορα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 228. Η 227 έχει καταπέσει. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12-12. Γι' αυτό και δεν είδα πλειοψηφία να υπάρχει. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά πάμε στη 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 243 έχουμε, είναι στη συμβαστική 28 που ψηφίσαμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα κατευθείαν στην 246. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 29, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε κατευθείαν στην 249, η ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 254. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 256. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 257. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 30. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 31 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πρέπει να πάμε στην 265 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 268 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 275 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 278 καταπίπτει και 279 καταπίπτει. Πάμε κατευθείαν στην, στην συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 282. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αυτήν πρέπει να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 282, 282. Πέρας της ψηφοφορίας. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 13 283 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 284 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 285 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ κατά αποχές εγκρί. 289 υπέρ α συγγνώμη 287 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 288 ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 291 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ κατά θα πρέπει να το ελέγξουμε. Ας επαληθεύσουμε για την 292. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13-12. 303. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296 προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Ας το επαληθεύσουμε. Πέρας. 297. 297 λοιπόν ε, είναι συμβατή, είναι ίδια, ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 υπέρ κατά πρέπει να τσεκάρουμε την 300 The vote Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 13 με 12. Συμβιβαστική 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 προφορική τροπολογία υπάρχει ένσταση όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 307 να την ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 307 πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 15 προς 7, 308. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 προς 6. Συμβιβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 310. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 310. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 310. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε την 310. Close the vote. Πέρας. 13 προς 12. Απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 313 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 314 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315 Σαφώς εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξετε. Ωραία, λοιπόν, 314 να κάνουμε έλεγχο. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. We close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. It's adopted, not clearly. Εγκρίνεται, όχι καθαρά, αλλά εγκρίνεται. 315. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 316 υπέρ κατά να ελέγξουμε δεν είναι πολύ σαφές άρχεται η ψηφοφορία πέγας εγκρίνεται 317 καταπίπτει 318 υπέρ Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται να ελέγξουμε. Ε, open the vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πρέπει να τα ελέγχουμε 319. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 προς 12. 320 υπέρ κατά να ελέγξουμε απορρίπτεται νομίζω αλλά ανοίγουμε την ψηφοφορία για την 320 πέρας Απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 321. Πέρας. Απορρίπτεται. 322 322 μάλλον να κάνουμε κατευθείαν ηλεκτρονική γιατί είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς. 322 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 323 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 324 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 325. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 326. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 327. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 328. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 329. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13 προ 11. 3-30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 331. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γιατί ήταν πολύ σαφής αυτή όλοι ψηφίζουν υπέρ. Ωραία, ας κάνουμε ε, left ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ευκολότερη. 331. Close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. 24 προς 0. 332. 332. Συγχαρητήρια στον Ολιβιέ. Δική σας ήταν τροπολογία. 332 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται καθαρά 333 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται σαφώς 330 4, 5, 6 έναρξη ψηφοφορίας λήξη απορρίπτεται 337 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 338 διανάτες χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 340 339 συγγνώμη 339 συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία ε, ε θα την κάνουμε ηλεκτρονικά γιατί είναι δύσκολη 339 άρχεται η ψηφοφορία Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Απορριπτέται σαφώς 3.40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 342 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 344 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.47 υπέρ απορρίφθηκε 3.47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.48 υπέρ κατά απορρίπτεται 348. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 349. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για το δεύτερο ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το τρίτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 350 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 351. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 352. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.55 καταπίπτει 3.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 358 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για την 360 Πέρας. Εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 362 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ κατά εγκρίνεται 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 366 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 372 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 375 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.79 υπέρ κατά Ας το ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία η 3.79 ελέγχεται αυτή τη στιγμή πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 380 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 381 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 382 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 383 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 384 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 385 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 ναι να ελέγξουμε την 387 Open the Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 15 388 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 393 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 394 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 395 394 μάλλον επαληθεύουμε το 394 άρχεται η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15-10. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν εδώ ε, αντιρρήσεις. Όχι. Ποιος είναι υπέρ. 395 έτσι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 397 υπέρ έχετε κάποιο ερώτημα 397 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται 398 προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 401 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 403 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 405 υπέρ κατά 405 θα πρέπει να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 406 με προφορική τροπολογία υπάρχει κάποια αντίρρηση όχι υπέρ κα, υπέρ κατά αποχές ε, Ας το επαληθεύσουμε. 406. Άχτη ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 407. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Άχτη ψηφοφορία, λέει ξανά η πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 408 άρχιδη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 409 υπέρ κατά εγκρίνεται 410 υπέρ κατά 410 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 411. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 412. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρχεται η ψηφοφορία 413 υπέρ κατά εγκρίνεται 414 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 415 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 416 υπέρ κατά Δεν είναι σαφή τα πράγματα. 416 πρέπει να το παληθεύσουμε. αρχεται Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 12-12. 417. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 418. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 419 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 421 υπέρ κατά πρέπει να το επαληθεύσουμε το 421 421 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται σαφώς. 4.22 με προφορική τροπολογία. Ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 423 δεν ψηφίζουμε, 424 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 425 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 427 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 427 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 428. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 429. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 430. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 431. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 432 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 436 τώρα υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ 4.36 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 4.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.40 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται 5 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 της ΑΦΕΤ εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία το πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα τροπολογίες από την Επιτροπή ΔΕΒΕ 7 υπέρ Θέλετε την ΑΦΕΤ 10 να την ελέγξουμε, μάλιστα. Εντάξει. Τροπολογία τη ΑΦΕΤ υπαρθμών 10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται σαφέστατα. ΔΕΒΕ 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και τώρα Επιτροπή Απασχόλησης, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Τροπολογία παρθων 5 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 της ΕΜΠΛ υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 19 ε, λέει τώρα η ομιλήτρια υπέρ κατά θα πρέπει να το επαληθεύσουμε για την 18 για την 18 λέει τώρα η πρόεδρος πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ, 18 ε, απορρίφθηκε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε, 20 της Επιτροπής Επασχόλησης, άρχιε ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά μάλλον απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά απορρίπτεται 31 υπέρ κατά εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε τώρα στις ε, τροπολογίες της NV 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV όχι NV 4 υπέρ κατά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 αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Τραν. Τραν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε όμως τροπολογία 4 της Τραν υπέρ. Ε, μάλλον άσχερη ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται όντως. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά θα πρέπει να το επαληθεύσουμε τραν 12 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 εκτός πεδίου. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 δεν ψηφίζουμε τώρα Επιτροπή Ρέγγι 2 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 της Επιτροπής Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ξεχωριστή ψηφοφορία τώρα. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. Γιατί ρέγγι 8. Πρώτο κομμάτι. Πρώτο σκέλος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Τώρα, περνάμε στην τροπολογίες της Επιτροπής Άγκρη. 6 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε. Παρακαλώ την Άγκρη 6 τσεκάρουμε. Απορρίπτεται. Άγκρη 11 τώρα. Εδώ έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε επί του πρώτου κομματιού. Υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο σκέλος του άγκρι, της τροπολογίας άγκρι 11. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται δεύτερο μέρος τώρα του 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές να το τσεκάρουμε όμως 11 λοιπόν ψηφίζουμε επί της 11 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 16-12 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις τροπολογίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Τέσσερα πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ κατά πρέπει να επαληθεύσουμε νομίζω την τροπολογία 6 της ΛΥΜΠΕ ψηφίζουμε Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 14-11. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα Επιτροπή Γυναικών. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά θέλετε να τσεκάρουμε το 9 μάλιστα να το τσεκάρουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 16-12 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά δεν είναι σαφές να το τσεκάρουμε να το τσεκάρουμε όλα μάλιστα 11 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 15 άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και τώρα έχουμε τελική ψηφοφορία ονομαστική ψηφοφορία για, το, για την πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Yes, I think we need five minutes to go to the bathroom for everybody. Πέντε λεπτά τεχνικό διάλειμμα οπωσδήποτε νομίζω για όλους. <laughs> Ελπίζω να ευχαριστήθηκατε τώρα το διάλειμμα όλοι. alles gut. Ich setze mich wieder Λοιπόν, πρέπει να βρω τώρα στα χαρτιά μου τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το σημείο 5, η απαλλαγή 2018 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συγγετριά μας είναι η Μαρία Καπίνη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρία για να ξεκινήσουμε πριν από τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, γραμματεία για την ε, εργασία αυτή που έγινε, τον σκιώδη τη βέβαια, αλλά και την γραμματεία που εργάστηκαν πολύ σκληρά. Εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα ε, κατά τη σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης. Ε, συναντήθηκα με τον Γενικό Διευθυντή, με τους σκιώδεις συγητές και με τη Γραμματεία και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς ακόμα μια φορά, καθώς και τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και προσπάθησαν να βελτιώσουν την έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω και για όλη τη δραστηριότητα το Κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την ε, εισηγήτρια και τους εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει και για την ομαδική τους εργασία, την ομαδική προσπάθεια και όλους όσους τους υποστήριξαν, καθώς και τη γραμματεία. Σας ευχαριστούμε όλους. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με την ψηφοφορία και ξεκινάω με την ψηφοφορία για το αν θα δώσουμε επαλλαγή ή όχι. Μιλάμε για ονομαστική τώρα ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. I... Πέρας. Uh, 21... 21 προς 1 και 3 αποχές. Τώρα, ερχόμαστε στην τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 16 ψήφους. Μετά. Συμβιβαστική πρόταση 2. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 8 του συναδέλφου Ομαριέ τέλος της ψηφοφορίας 13-13 απορρίπτεται 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 10 υπέρ. Α, συγγνώμη. Έχει καταπέσει. Ε, 11 υπέρ κατά. Ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την επαλήθευση για τροπολογία 11. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Μετά Έχουμε το αρχικό κείμενο της εισηγήτριας. Ah, if Αν θέλετε να διαγραφεί η παράγραφος αυτή, ψηφίζετε αρνητικά. Αν δεν θέλετε να διαγραφεί, ψηφίζετε θετικά. Για να διαγραφή πρέπει να ψηφίσετε μείον. Για να παραμείνει η παράγραφος να ψηφίσετε συν. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία εννοώ. Ποιος θέλει, όποιος θέλει να διαγραφεί θα ψηφίσει μείον και όποιος θέλει να παραμείνει θα ψηφίσει συν. Άρχεται η ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 23. πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 15-11. Επόμενη τροπολογία. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές για την τροπολογία 12. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Μετά, παρα, ε, τροπολογία 13. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 15. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Κατά. Εγκρίνεται. Μπορούμε να το επαληθεύσουμε, αλλά νομίζω ότι εγκρίθηκε. Mm Για το δεύτερο τμήμα. Διανατάσεως της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 3. Ψήφι υπέρ, κατά, ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ανοιχτή η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Τώρα έχει λήξει. Κάποιοι συνάδελφοι χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο. Εγκρίνεται 14-8. Είναι το αποτέλεσμα. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 4. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is still open on compromise for, Somebody that's not vote? Okay. Okay, now. Λοιπόν, πέρασε τη ψηφοφορία τώρα. Απορρίπτεται. Τώρα, πρέπει να ψηφίσουμε την 22 νομίζω. Σωστά. 22 και 23. Ε, πρώτα 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και γίνεται η επαλήθευση για την τροπολογία 24. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 14-12. 25 ε, λοιπόν και 26 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει και πάλι να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα, τις επαληθεύσουμε και πάλι. Μου φαίνεται θα τις επαληθεύσουμε όλες έτσι όπως πάμε. Για την 27 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Καταπίπτει. Η 29 καταπίπτει. Έχετε δίκιο. 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Ψήφι υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Επαλήθευση. Ας το επαληθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να δείχνετε πιο καλά, πιο καθαρά τι ψηφίζετε. 37. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. Γιατί ψήφισε και η Ρινιού. Λοιπόν, 37 ε, επαληθεύουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την 45 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις 47. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 13-11. 48. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 ψήφι υπέρ, κατά, ας το επαληθεύσουμε. 49. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15-11. Ε, τροπολογία 50. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας το επαληθεύσουμε για την 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 τώρα πάμε. Α, όχι, συγγνώμη, 61. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Τέσσερις ομάδες ψήφισαν υπέρ. Μπορούμε να το επαληθεύσουμε αν θέλετε. Για την 62 δεν υπάρχει πρόβλημα να επαληθεύσουμε. 62 λοιπόν, τροπολογία 62. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, κυριακούς, πέρας της ψηφοφορίας. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 καταπίπτει 67 αποσύρθηκε 68 υπέρ Κατά. Σας παρακαλώ, σηκώνετε τα χέρια σας. Νομίζω ότι απορρίπτεται η 69. 69. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να το επαληθεύσουμε. Επαλήθευση για την τροπολογία 69. Πέρας της ψηφοφορίας. 15-12 απορρίπτεται. 70 ψήφι υπέρ. Κατά. Σαφώς απορρίπτεται. 71 και 72. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 71 και 72. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 73 και 74 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 73 και 74. Πέρας της ψηφοφορίας. 75. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 76 ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 76? Μάλιστα. Ας το κάνουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εβδομήντα εφτά. Η εβδομήντα εννιά, καταπίπτει. Καταπίπτει λέει αν εβδομήντα εφτά. Αν η 75 εγκριθεί. Την 75 την εγκρίναμε. Όχι, την 76 λέει εκεί. Μάλιστα. Ψηφίζουμε για την 77. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78. Καταπίπτει. 79. Πρέπει να ψηφίσουμε για την 79. Ψήφι υπέρ. Κατά. Όχι, δεν καταπίπτει. Για την 79 σας παρακαλώ, άλλη μια φορά. Ψήφι υπέρ για την 79. Κατά. Το ΕΛΚ δεν έχει δείξει πώς ψηφίζει. Ας την επαληθεύσουμε, την 79. Γιατί αν κανείς δεν σηκώνει το χέρι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Εγκρίνεται. Σαφώς. 81. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αλλά δεν βλέπω εδώ στο κέντρο τι κάνουν. Επαληθεύουμε για την 82. I think it's adopted, but uh, we the vote. Yes, it's σαφώς εγκρίνεται. 83. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε νομίζω. Yes, uh, we, but you have to vote now. <laughs> Uh, uh, we close the vote. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. 84 ψήφι υπέρ. Κατά. Εκρίνεται. 85, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. εγκρίνεται 88 υπέρ κατά θα μπορούσε σας παρακαλώ το έλκυ να ψηφίζει γιατί έχουμε πρόβλημα αν δεν ψηφίζετε τι ψηφίζετε υπέρ ή κατά ας ξαναψηφίσουμε ποιος είναι υπέρ κατά νομίζω ότι είναι κοντά ε, πρέπει να το επαληθεύσουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Είστε σίγουροι. Απορρίπτεται. 12-12. 89. Να μια καλή τροπολογία γιατί είμαι και εγώ συντάκτρια. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 90. Ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται 91 ψήφι υπέρ ψήφι κατά εγκρίνεται 92 υπέρ κατά πρέπει να το επαληθεύσουμε γιατί κάποιοι δεν ψηφίζουν Πέραση τη ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 93. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 94. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. Σαφώς ε, ε, εγκρίνεται. 95. Ψήφι υπέρ κατά εδώ πρέπει να το επαληθεύσουμε πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 96 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει καμία αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν για την προφορική αυτή τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα πάνω στο πρωτότυπο κείμενο. Ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου. κατά απορρίπτεται. Μετά 98 υπέρ κατά εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά εγκρίνεται. 100 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Για την 100 μιλάμε τώρα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι κατά. Α, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Η 100 καταπίπτει. Ε, η 101 έχει αποσυρθεί. Η 102. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Για την 102. 102 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είχαμε αποχή και τα υπόλοιπα ήταν συν. Με την αποχή μπορούμε να το ελέγξουμε. Εντάξει, το ελέγξουμε για να το δείξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 23 εναντί μίας και μίας εποχής. 105 έχει αποσύρθει 106 καταπίπτει αφού πρέπει να ψηφίσουμε την 104. Ποιος είναι υπέρ. 104 ψηφίσουμε την 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 106. Υπέρ. Δεν ψηφίσαμε την 105, όχι. Έχει αποσυρθεί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 με προφορική τροπολογία. Ε, ενστάσεις. Πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 109. Πιο υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. We please vote on Να ψηφίσουμε την 109. Ε, Απορρίπτεται. 14-14. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ καταπίπτει συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε νομίζω ας ελέγξουμε την 131 Πέρας. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 138. Πέρας. Απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται. Μπορούμε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε 140. Πέρας. Απορρίπτεται 14-14. Δεν ε, το έβλεπα καλά. 141. Δεν φαινόταν ε, καλά.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 Προφορική τροπολογία για την 146 έναρξη πέρας εγκρίνεται. Μπορούμε να πάμε στην 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε τώρα για την 150 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 13. Δεν υπάρχει πρόβλημα. closed. I'm in favor. It's rejected. Απορρίπτεται. 150. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 100. Να το ελέγξουμε 150. Ελέγχουμε την 150. Πέρας. Εγκρίνεται. 153. Καταπίπτει. 149. Καταπίπτει. 151. Ίδια με την 13. 151 πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Μετά από 600 τροπολογίας 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 με ονομαστική ψηφοφορία 16 υπέρ άρχεται ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία για την συμβιβαστική 16 πέρας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 14 προς 13, 176 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 176. Το ίδιο, 14-13, 177, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, η ίδια νομίζω είναι. 14-13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 177. Είστε υπέρ. Πέρας ψηφοφορια 14 προς 13. Εγκρίνεται. Πάμε στην 178. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 14-13 νομίζω είναι. Ας το τσεκάρουμε. δεν είδα τον Ολίβια. Συγγνώμη. Απορρίπτεται. Αλλά ας κάνουμε την ψηφοφορία 178. Άρχεται η ψηφοφορία. για την 178 πέρας απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά να το ελέγξουμε αλλά νομίζω ότι εγκρινέται ψηφίζουμε για την 183 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 181

υπέρ κατά εγκρίνεται 186 υπέρ 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε 193 εγκρίνεται Συμβιβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 195 πέρας εγκρίνεται 196 υπέρ κατά εγκρίνεται 197 υπέρ κατά εγκρίνεται νομίζω να ελέγξουμε αλλά νομίζω ότι εγκρίνεται 197 14-13 κάτι τέτοιο ε, πέρας όχι απορρίπτεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά να ελέγξουμε πέρας ελέγχου απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 199 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Close. Πέρας εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω 201 υπέρ κατά εγκρίνεται να το ελέγξουμε Πέρας. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 22. 22. υπέρ Συμβεστική 22 υπέρ κατά εγκρινέται 207 υπέρ κατά εγκρίνεται η συμβεστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία και ψηφοφορία σε τμήματα. Ας ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα με την προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση. Υπάρχει ένσταση. Οπότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου. Κατά απορρίπτεται. Όταν έχουμε ε, τώρα 214 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε ξανά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 214. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματο στο σύνολό τη. Όπω τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω ότι έχετε τεράστια πλειοψηφία. 24. Μπράβο. Θέλει κάποιος να κάνουμε διάλειμμα. Όχι. Κύριε Νόβακοφ, πρέπει να ψηφίσετε. Μαρινέσκου. Α, ο Μαρινέσκου θα ψηφίσει. Please. Παρακαλώ, μην σηκώνεστε. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. Γεια σας, καλημέρα. Πρώτα ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Α, πρώτα απ' όλα η συγγήτρια. Ήθελε το λόγο η κυρία Ριβαζή. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Στην ημερήσια διάταξη σημείο 6. Το σημείο 6. Απαλλαγή 2018. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 10ο και 11 ετά. Η συγκήτρια κυρία Ριβάζη και ο συνάδελφος Φρόντε έχει δίκιο βιάστηκα υπερβολικά καθώς η συγκήτρια δεν είναι εδώ δεν μπορεί να πάρει το λόγο αυτή τη στιγμή θα ήθελε κάποιος από τους πρασίνους να πει κάτι όχι δεν θέλει να την καθιστήσει κανείς ε, ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία λοιπόν ποιος είναι υπέρ ποιος είναι κατά απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά απορρίπτεται μετά έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία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 κατά να το ελέγξουμε We check number 9. Τροπολογία 9 λοιπόν, επαλήθευση. It's 40... Πέρα ψηφοφορίας 14-8 Τροπολογία 10 υπέρ κατά νομίζω ότι το ίδιο θα βγει και εδώ εγκρίνεται θέλετε να το τσεκάρουμε μάλιστα τροπολογία 10 ψηφίζουμε λοιπόν επαλήθευση Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 14-8. 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το τσεκάρουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Νομίζω ήταν σαφής η πλειοψηφία. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο σκέλος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο σκέλος. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο σκέλος τώρα. Με τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Ναι, ναι. Έχετε κάποια αντίρρηση. Είστε κατά της προφορικής τροπολογίας, μάλιστα. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν επί του αρχικού κειμένου. Ποιο είναι υπέρ. Δεν ακούμε τον ομιλητή εκτό μικροφώνου. είναι καλούμε την Κομισιόν να... Αυτό λέει το κείμενο. Να σταματήσει ε, την, ε, να ακυρώσει τα τουλάχιστον εκατομμύρια που έχουν διατεθεί για την Ερυθρέα και τα λοιπά. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί του αρχικού κειμένου, λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Κομισιόν δεν θα παραδίδει μηχανήματα, εξοπλισμό. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί του αρχικού κειμένου. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Δεύτερο κομμάτι, έτσι. Δεύτερο σκέλος της ε, τροπολογίας 41, ε, παράγραφος 68. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 42 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43, 44 εδώ έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, υπάρχει μάλλον προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ε, μάλλον δεν το δέχεται ο συνάδελφος. Ζητούμε από την Κομισιόν να εξετάσει την ακύρωση ε, την ε, οικονομική υποστήριξη κτλ. Μάλιστα, ψηφίσουμε το αρχικού κειμένου λοιπόν, υπέρ. Να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τελική ψηφοφορία ονομαστική επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Because we stop it. Yeah. Είναι 21... 21 υπέρ, μια κατά δύο εποχές. En español. We continue the... Συνεχίζουμε στις 3 την ψηφοφορία. Close the session. By now. Πέρα τη συνεδρίαση ε, για το πρωί. Not closing. Not closing. Όχι, όχι, δεν ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Ναι, συγγνώμη, υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Ο άλφος Μαρινέσκου θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα για την Όλαφ. Τώρα το θυμήθηκα. Υπάρχει άλλο ένα σημείο. Όχι για την Όλαφ σίγουρα. So, so we had several uh, technical Λοιπόν, είχαμε μια σειρά από τεχνικέ συναντήσει, μόνο έναν τρίλογο. Προβλέπεται επίση 18 Μαρτίου τρίλογο, τριμερή διάλογο. Έχω λάβει κάποια μηνύματα από διάφορε πολιτικέ ομάδε που θέλουν να ε, εργαστούν μόνο αφού ε, ψηφιστεί η απαλλαγή. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γι' αυτό και ετοίμασα κάποια αριθμητικά στοιχεία εδώ για να είμαι σαφής. Αυτός ο κανονισμός βασίζεται ε, εν μέρη σε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιπλέον το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες που σχετίζονται με την Όλαφ. όχι με τη συνεδρία, στη συνεργασία μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για το πρώτο σκέλο, λοιπόν, την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν 77 παράγραφοι, α πούμε. Οι 56 είναι αντικείμενο συμφωνία. 8, 8, για 8 υπάρχουν σημαντικές διαφορές, ε, σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και Οικονομικών και Συμβουλίου και 11 είναι αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 32 είναι συμφωνημένες, 5 παρουσιάζουν δυσκολίες και ε, υπάρχουν ακόμα 13 που είναι υπό διαπραγμάτευση. Και υπάρχουν ακόμα και τρει ε, τροπολογίε από το Συμβούλιο που είναι προ συζήτηση. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν τροπολογίες ε, που έχουν σημα... παρουσιάζουν σημαντικά στοιχεία, ΦΠΑ, τραπεζικοί λογαριασμοί. Ε, ε, όμως, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, έχουν να κάνουν κυρίως με την έκθεση, την αναφορά δηλαδή που θα πρέπει να δίνει η Όλαφ προς το Κοινοβούλιο. Ενημέρωση, συνεργασία, μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν είναι τόσο περίπλοκα όλα αυτά. Αυτό που είναι περίπλοκο είναι ότι εγώ ή εμείς διαπραγματευόμαστε ως Κοινοβούλιο όχι με το Συμβούλιο αλλά με την Όλαφ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Διότι κάθε φορά που το, το Συμβούλιο ρωτάει την Κομισιόν και στην Κομισιόν, γιατί για την Κομισιόν απαντάει η Όλαφ. Και μας είπαν σαφώς ότι έχουν οι ίδιοι, η όλα, δηλαδή, έχει εντολή διαπραγμάτευση. Προσπάθησα εγώ να εξηγήσω ότι εγώ διαπραγματεύομαι με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι εκεί ω παρατηρητή. Και μα είπαν όχι. Εδώ έχουμε τριμερή διάλογο, έχω λάβει εντολή διαπραγμάτευση. Πρώτη φορά το ακούω και αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι η Όλαφ δεν θέλει να λάβει αυτές τις υποχρεώσεις να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ή να συζητάει με, το, με την, ε, για το Γενικό Εισαγγελέα ή ε, το να καλείται ο Γενικός Εισαγγελέας παραδείγματος χάρη ε, στην αντίσια συνάντηση με το Συμβούλιο, την Κομισιόν δηλαδή δεν θέλουν ο Γενικό Εισαγγελέας να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Γενικό Γραμματέα. Και αυτά τα λέει η Όλαφ, έτσι, όχι το Συμβούλιο η Αυτό είναι ένα παράδειγμα που σας δίνω. Το πρόβλημα επίσης έχει να κάνει με τον έλεγχο. Την πρόταση του Κοινοβουλίου. Εγώ επέβαλα μια άλλη πρόταση που γίνεται αποδεκτή από την Εποπτική Αρχή, την Εποπτική Επιτροπή, και η έκπληξη για μένα ήταν ότι η Όλαφ υποστηρίζει την πρώτη πρόταση του Κοινοβουλίου, την προηγούμενη. Γιατί, διότι αυτή ήταν η πρόταση τη Κομισιόν πριν από μερικά χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί το κάνουν αυτό επειδή είναι πιο δύσκολο να το δεχτεί το Συμβούλιο, βέβαια. Η πρότασή μου είναι να δώσουμε τα ίδια καθήκοντα σε κάποιον αλλά εντό της εποπτικής αυτή τη Επιτροπής, διότι κάνουν το ίδιο πράγμα. Παρακολουθούν τις ε, διαδικαστικές εγγύησει Και αυτοί οι ελεγκτές και ε, η υποπτική Επιτροπή. Η Εποπτική Επιτροπή εξ των και ε, ο ελεγκτής κατά τη διάρκεια της έρευνας. γιατί να μην το κάνει αυτό η ίδια οντότητα αφού κάνουν το ίδιο πράγμα. Αυτά κυρίως Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για μια τροπολογία του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη που δίνω αυτά τα παραδείγματα, αλλά έτσι είναι. Το Κοινοβούλιο προτείνει ο Γενικός Διευθυντής να μην διενεργεί ο ίδιος μια έρευνα. Γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι αφαιρούμε το δικαίωμα του Γενικού Διευθυντή, εν πάση περιπτώσει. Ο Γενικός Διευθυντής βεβαίως και ασκεί τα καθήκοντά του και καθοδηγεί όλες τις έρευνες. Αλλά δεν την κάνει ο ίδιος την έρευνα. Αυτό ζητάει το Κοινοβούλιο. Όχι όμως, λέει η Όλαφ, ούτε η Όλαφ το δέχεται, ούτε και το Συμβούλιο. Αυτά. Εγώ δέθηκα κάποιες εξορτάσεις ε, του Συμβουλίου μια παρατυπία που υπήρχε σε κάποια άλλη τροπολογία του Κοινοβουλίου ε, μάλλον ο ορισμός της παρατυπίας του irregularity έχει τροποποιηθεί και βεβαίως το θέμα των εσωτερικών και των εξωτερικών ερευνών ε, ήταν μια καλή ιδέα αυτή να αλλάξει η ονομασία ο τίτλος της έρευνας, όμως ε, είναι πολλά άλλα έγγραφα που θα πρέπει να τροποποιηθούν στην περίπτωση αυτή. Το περιεχόμενο λοιπόν είναι αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο, όμως το όνομα, ο τίτλος της έρευνας ε, μένει ως είχε, εσωτερική και εξωτερική δηλαδή. Αυτά από μένα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου ε, για την πολύτιμη εργασία. Σας ξέρουμε ότι είναι περίπλοκο αυτό που έχετε να κάνετε. Ματίνα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Είχαμε, είχαμε τεχνικές συναντήσεις και συμφωνήσαμε ότι θα το συζητήσουμε αυτό στις συναντήσεις των σκιωδών εισογητών. Οπότε παρακαλώ να γίνει μια συνεδρία σκηνοδών εισογητών και να συζητηθεί αυτή η πρόταση, διότι εδώ δίνεται η εντύπωση ότι ε, δεν ακολουθούμε την εντολή που λάβαμε μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και πρέπει να το συζητήσουμε. Η απόφαση ήταν να μην το αφήσουμε αυτό σε τεχνικό επίπεδο. Δεν δηλαδή, να κάνει το προσωπικό μα εκεί, διότι δεν μπορούμε να είμαστε και σε δύο μέρη ταυτόχρονα, όταν λαμβάνει η χώρα συνέντευξη τη Επιτροπή και να έχουμε και τεχνική συνάντηση. Α γίνει λοιπόν συνέντευξη των σχεδόν εισαγητών για να το δούμε. Ε, ευχαριστώ για το έργο σα. Ευχαρίστω, λέει ο κ. Μαρινέσκου. Εγώ δεν, σε καμιά περίπτωση πάντω δεν παρέκλεινα από την εντολή. Και ό,τι έκανα, και πρέπει να το ξέρετε βέβαια, διότι η βοηθή σας, η συμβουλή σας ήταν εκεί. Ε, εσείς δεν ήσασταν. Ήταν, ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής μας. Ακούστε, εγώ προτείνω, πρότεινα 12 Μαρτίου συνέδρια στους κοινωνικούς αγητών. Δεν έχω λάβει απάντηση από κανέναν. Η μόνη απάντηση είναι ότι θέλετε να εργαστείτε μετά την ολοκλήρωση της απαλλαγής. Αυτό όμως είναι μετά τις 18 Μαρτίου και η Κροατική Προεδρία η οποία θέλει να εργαστεί, θέλει να προχωρήσει, έτσι, είναι εξαιρετικά συνεργάσιμη. 18 Μαρτίου προτείνουν. Να κάνω μια πρόταση πριν να αναστατωθεί και τσεκωθεί οποιοδήποτε. Θα θέλαμε να υπάρχει μια στάση από κάθε ομάδα. Ε, ξέρουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα, είναι μεγάλο ο φόρτο. Το ίδιο συμβαίνει και για τον κύριο Μαρινέσκο, Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ε, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να συζητήσουμε. Υπάρχει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει καμία κακή βούληση από καμία πλευρά. Υπάρχει τεράστια πίεση όταν είσαι μόνος σου ε, και έχεις αυτές τις 2.000 ε, τροπολογίες ε, σας θαυμάζω για αυτά που έχετε κάνει απ' την άλλη όμως πρέπει να συνεχίσει και ο συνάδελφος ο κ. Μαρινάσκου που λίγο Αμοιβέ εμπιστοσύνη βάσει των όσων ψηφίσαμε μπορούμε να διαπραγματευτούμε και μετά αν προκύψει κάτι νέο τώρα η απαλλαγή έχει δοθεί θα δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση των σκηνιωδών και ελπίζω να πάνε όλα καλά λίγο κατανόηση και από τις δύο πλευρές και μετά στην επόμενη και εδώ μπορείτε να το συζητήσετε όλα αυτά να πάνε όλα καλά αλλά δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε όλα θα έδινε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση αυτό να μην γίνει κανένα τρίλογο ε, παρότι το επιθυμούν οι Κροάτε. Ε, και τώρα οι Κροάτε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση όλοι οπότε θέλω να ευχαριστήσω και τους Κιώδης ε, που δεσμεύτηκαν θα μπορούσατε ενδεχομένω στην επόμενη συνάντηση να τα καταφέρετε. Είναι δύσκολη εργασία και προσπαθεί και ο δικό μα συγκεκριτή να υπερασπιστεί τα δικά μα ενδιαφέρον, αυτά που μα ενδιαφέρουν εμά. Δεν είναι εύκολο φυσικά με το Συμβούλιο και την Κομισιόν μαζί, αλλά α κάνουμε ό,τι μπορούμε. Για τη συνάντηση των σκιωδιωδών ε, έχουμε στις 12 Μαρτίου. Μια εβδομάδα δηλαδή πριν ε, τον τριλόγο. Ζήτησε η Πρόεδρος ε, σεβασμό. Εμείς έχουμε μόνο ένα σύμβουλο, σεβαστείτε το. Δεν μπορούμε να είμαστε παντού ταυτόχρονα, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε έναν άνθρωπο στα δύο ή στα τρία. Θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Μετά την απαλλαγή λοιπόν. Δεν θέλω να πω τώρα στα ζητήματα περιεχομένου, διότι θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε, διότι δεν έχετε δίκιο στα που λέτε. Ας το κάνουμε στις συνεδρίες των σκηνών εισαγητών τι είπατε, δεν εξήγησα σωστά αυτά που είπα. Συγγνώμη, ήδη εδώ μπαίνει θέμα σεβασμού, έτσι. Οπότε σεβαστείτε με, έτσι. Εγώ λέω μόνο αυτά που συμβαίνουν. Γνωρίζω το φάκελο. Πολύ καλά. Μην κοιτάζετε τους συμβούλους σας. Εμένα να κοιτάτε. Γνωρίζω το φάκελο. Αυτό που είπα είναι αλήθεια. Θα πρότεινε αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει δυσπιστία από αμφότερε πλευρέ. Ο Μαριάν θα πρέπει να συνεχίσει και εσύ, Μαρτίνα, αν βρει κάτι από πλευρά σου, σε παρακαλώ να κάνει ένα ραντεβού πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαριάν για να εξηγήσει που ενδεχομένω υπάρχει κάποια παρανόηση και έτσι πιστεύω θα λυθεί η παρανόηση αυτή, η παραξήγηση αυτή που υπάρχει. Ε, ε, και να ακολουθήσουμε και αυτά που φασίστηκαν εδώ φυσικά ο, ο κύριος Φλάναγκαν. Έχουμε περάσει στον κόσμο των κακών τρόπων. Δεν μπορεί ο καθένας να συμπεριφέρεται. Όλο ο κόσμο μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Δεν μπορείτε να απαιτείτε εσείς κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εδώ είναι το έκτο μου, η έκτη μου χρονιά. Ουδέποτε έχω ακούσει κάτι που να χαρακτηρίζεται από τόση ε, άγνοια ε, από όσο αυτό που είπατε και θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Σα παρακολουθώ. Αυτή τη στιγμή μην επιτίθεστε ο ένας στον άλλο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο όπως είπα, είναι μεγάλες. Υπάρχει πίεση από την κρατική προεδρία και εμεί θέλουμε το αρχείο αυτό από την... Ε, Ω κοινοβούλιο θέλουμε να ενδυναμωθεί ε, η Όλαφ, αλλά δεν μπορεί να αποφασιστεί αυτό χωρίς να γίνει μια καλή συζήτηση στην ε, συνάντηση των σκιωδών. Θα πρέπει να συμφωνηθούν κάποια πράγματα εκεί. Οπότε δείξτε λίγη εμπιστοσύνη μέχρι τον επόμενο τρίλογο. Ε, ξέρεις πότε θα γίνει Μαριάν. 18 Μαρτίου. Προτείνω 12 Μαρτίου εγώ. Αν έχω απαντήσει στα χέρια μου, προτείνω 12 Μαρτίου. Γιατί για μένα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στο Στρασβούργο είναι εντάξει. Όποια μέρα θέλετε. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί τουλάχιστον, Μαριάννα, θα μπορούσε να περιορίσεις λίγο, να γνωρίζουμε ακριβώς πότε, ακριβώς 18 για παράδειγμα, αν θα συζητήσουμε ολόκληρο το αρχείο, ένα, δύο συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα συζητηθούν εκείνη τη μέρα. Ξέρεις ακριβώς τι θα συζητηθεί ήδη. Ξέρεις τι θα συζητήσετε στις 18, ποιο σημείο. Όχι. Δεν έχω κάτι στην ατζέντα αυτή τη στιγμή, αλλά θα συζητήσουμε και θα την καθορίσουμε φυσικά. Έτσι κάναμε μαζί, έτσι κάνουμε ανέκαθεν. Τι ατζέντε και των τεχνικών συναντήσεων και του πρωτού τριλόγου. Όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο φυσικά να συζητηθεί όλο το αρχείο Όλαφ. Ε, δεν μπορούμε να τον μπλοκάρουμε, όπω καταλαβαίνετε, όλο το αρχείο. Γι' αυτό θα έλεγα, αν υπάρχουν ερωτήσεις από ευρωβουλευτές, ε, παρακαλώ, ελάτε σε επαφή με τον Μαριάν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και θα συνεχιστούν και μετά την απαλλαγή. Δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό συνεδρία των συντονιστών αύριο. Και να προσπαθούμε να είμαστε και ευγενικοί, έτσι, όταν μιλάμε μεταξύ μας. Είναι στην εμείς διάταξη. But then you have to know at the end, if we are talking at the coordinators, I hadn't seen this point. Ακούστε, αν το δούμε στις συντονιστές πάντως πρέπει να σας πω ότι η Κροατική Προεδρία και το Συμβούλιο θα πούν το Κοινοβούλιο θέλει να σταματήσει την Όλαφ. Περιμένουμε το Κοινοβούλιο. Σας το λέω σαφώς. Αυτό θα μας πούν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε αύριο συντονιστέ. Δεν ξέρω, Μάρια, αν θα έχει χρόνο, αν θα είσαι εκεί αύριο το πρωί. Μάλιστα, θα το κάνω εγώ τότε. Πες το και στον Τόμα Σεντόφσκι. Ο συντονιστής του ΕΛΚ μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα στους άλλους συντονιστές. Θα ήταν πρόβλημα να πάμε τον όλα δύο-τρεις μήνες πίσω. Πολύ ωραίο. Δύο και μισή υπάρχει συνάντηση για την αποστολή στην Τσεχία και στις τρεις συνεχίζουμε τις εργασίες μας εδώ και συνεχίζουμε τις, με τις Ευχαριστώ Μάρια, σας ευχαριστώ όλους.